χρειαστεί ενός λεπτού σιγή τώρα για αυτή την ιδιαίτερα μαχητική δημοσιογράφο αμήντορα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία. Μάλιστα κυρία Χάρμς. Θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβουλίο ότι ο πρόεδρος Μπούσεκ για αυτό ακριβώς το θέμα έκανε μια δημόσια δήλωση την οποία θα σας διαβάσω. Με μεγάλη λύπη έμαθα τον τραγικό θάνατο της Νατάλιας Δεμίροβα που είχε απαχθεί νωρίτερα σήμερα στον Κρόσνη. Εκ ξονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας ε, στην οικογένεια και τους φίλους ε, της αποθανούσας. Η Νατάλια Εσδεμίροβα ήταν μια ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και σημαντική ερευνήτρια για θέματα Τσετσενίας. Το 2005 είχε λάβει το ε, μετάλλιο Ρομπέρ Σουμάν από την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμούμε το έργο της ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πρόθεση ε, της, ε, του κράτους δικαίου και καλούμε τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ξεκινήσουν μια έρευνα σε βάθος για το θάνατό της και να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να δικαστούν οι πέτοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, βρίσκεται ε, μπροστά στο μέτωπο της υπεράσπισης της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας ε, σε όλους αυτούς που αγωνίζονται παντού στον κόσμο για τις ίδιες αρχές με αυτές της Νατάλια Εσδεμίροβα. Και τώρα κυρία Χάρμς. Η Προεδρία, κυρία Χάρμ, σύμφωνα με την πρότασή σας. Θα, διατηρήσουμε, θα τηρήσουμε ένα λεπτό σιγής προς τη μνήμη της. Κυρίε και κύριοι, εξαντλήσαμε τη μερίσια διάταξή μα. Τα πρακτικά θα σας υποβληθούν στην ε, επόμενη σύνοδο προς έγκριση. Διακόπτουμε. Κυρίως ότι λήξη συνεδρίασης.